E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι επιδοκιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύω στην Ολομέλεια. Πάμε στις ψηφοφορίε. Πρώτη έκθεση της κυρίας Πατρίτσια Σούλιν αφορά την απόφαση την πρόταση απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 τη Διοργανική Συμφωνία τη Δευτέρα Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία, τη Συνεργασία σε Δημοσιονομικά Θέματα και τη Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κτο ε, είναι e, Κατά. Ναι, ναι, ονομαστική κλίση, το είπαμε. Αποχές. Uh, Σα ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Έχουμε ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτείται εδώ πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, και εγκρίνεται η έκθεση της κυρίας Σούλη. Περνάμε στη δεύτερη έκθεση που είναι του κυρίου Ρούμπιχ. Αφορά την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 τη Διοργανική Συμφωνία τη Δευτέρα Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική επιθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και πάλι η ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, λέει ο Πρόεδρος. Kto z Państwa jest przeciwny? Kata. Kto z Państwa... Αποχές. E, głosowanie jest zamknięte. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εδώ απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία. Πάνω από τα τρία πέμπτα των, ψήφων, των ε, Ευρωβουλευτών έχουν ψηφίσει πληρούνται οι προϋποθέσεις, εγκρίνεται η έκθεση. Επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Πέτρη Σάρβαμα. Έκθεση Σάρβαμα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία.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 Εγκρίνεται η έκθεση του κυρίου Σάρβαμα και περνάμε στην τελευταία έκθεση της κυρίας Ιζαμπέλ Τομά. Αφορά κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το λόγο έχει η συγγήτρια, η κυρία Ιζαμπέλ Τομά, για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Φοβούμαι όμως ότι δεδομένη τη ατμόσφαιρας, εδώ δεν ξέρω τι τρέχει, ε, δύσκολο θα είναι στις 25 Απριλίου η ε, Γαλλία υπέβαλε ε, αίτηση για άντληση χρημάτων από το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση από, της εταιρείας ΠΕΣΑ από την πόλη ΡΕΝ και μια άλλη πόλη, 2.300 εργαζόμενοι ε, απολυμμένοι, δεν έχουν ξαναβρει δουλειά, είναι στην ανεργία. Το σχέδιο αυτό έχει καταρτιστεί για να τους βοηθήσει να βρουν ε, εργασία. Παρακαλώ να το εγκρίνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ.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 The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Ogłaszam wyniki. Głosowanie jest... Εγκρίνεται η έκθεση της κυρίας Διακοπή της Συνόδου μέχρι τις 3 και σας εύχομαι καλή όρεξη.